Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας λοιπόν. Καταρχάς θα ξεκινήσω με μία ανακοίνωση λόγω της εκένωσης ε, του κτηρίου που έγινε για λόγους δοκιμής σήμερα. Όλες οι επεξηγήσεις ψήφου στα θέματα τα οποία ψηφίστηκαν το πρωί θα γίνουν αύριο. Θα διευκρινιστούν όλα αυτά χρονικά λοιπόν. Αύριο επίσης θα ολοκληρώσουμε καιρός νομίζω τις ψηφοφορίες οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν σήμερα. Και οι ψηφοφορίες οι οποίες διακόπησαν θα συνεχιστούν αύριο. Δεν θα υπάρξει κάποια σημαντική διαφορά. Τα πρακτικά είναι διαθέσιμα, δεν βλέπω να υπάρχουν σχόλια θεωρούνται αποδεκτά. Το πρώτο θέμα λοιπόν το οποίο έχουμε στην ημερήσια διάταξη είναι η ώρα των ερωτήσεων με τον πρόεδρο της, της Επιτροπής. Η πρώτη ερώτηση θα τεθεί από τον κύριο Μάνφρεντ Βέμπα εξ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Κύριε Πρόεδρε, Λοιπόν, επιβιώσαμε τις διαδικασίες εκένωσης του κτηρίου. Ήταν μια διαδικασία που μας έκανε λίγο να χαμογελάσουμε. Ας θέσω λοιπόν τώρα τα ερωτήματά μου εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Βλέποντας τις τελευταίες μέρες τι συμβαίνει στην Μεσόγειο, όπου πολλοί φεύγουν από τη Βόρεια Αφρική για να έλθουν στην Νότια Ευρώπη, Κάποιοι δυστυχώς χάθηκαν στη θάλασσα. Το πρόβλημα είναι σοβαρότατο και θα πρέπει σε αυτό το δράμα να δώσουμε μια απάντηση. Εξ ονόματος λοιπόν του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ήθελα να ρωτήσω από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας πει τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι κάνει το Frontex, υπάρχουν επαρκείς πόροι στα πλαίσια του Frontex. Για επιτόπια δράση Ποια είναι η νομική βάση για τη δράση του Frontex εκεί. Και στις συζητήσεις που έχετε με τις χώρες προέλευσης, την Ισία, Αίγυπτο κτλ. Έχει υπάρξει πρόοδο σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Βέμπερ. Όλοι είδαμε τα τελευταία γεγονότα, τα οποία δυστυχώς οδήγησαν στην απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να αναλυφθεί περαιτέρω δράση. Υπήρξε οικονομική βοήθεια προς τις χώρες αυτές, οι οποίες η οικονομική βοήθεια ανήλθε σε 100 εκατομμύρια ευρώ, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει οι χώρες της Μεσογείου να συνεχίσουν τις προσπάθειες. Απαιτούνται να γίνουν περισσότερα. Η απάντησή μου λοιπόν προς εσάς είναι ότι πράγματι απαιτούνται περισσότεροι πόροι για το Frontex. Η πρόταση για την νομική βάση θα πρέπει να γίνει το ταχύτατο δέκτη και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δείξουν την πολιτική τους βούληση και την αλληλεγγύη θέτοντας στη διάθεση της Ένωσης τα μέσα τα οποία λείπουν. Για να υπάρξει κάτι τέτοιο απαιτείται φυσικά η συνεργασία όλων των κρατών μελών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεύτερη ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την παρουσίαση που κάνατε. Λέτε ότι προς το παρόν χρειαζόμαστε επιπλέον πόρους για το Frontex. Θέλω να ξέρω τα κράτη δεν ήταν επαρκώς διατεθειμένα να δώσουν τους επαρκείς πόρους στο Frontex. Έχουμε το κουτί με τα εργαλεία, αλλά φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν ε, να υποστηρίξουν τη Frontex. Αυτό πρέπει ίσως να το αλλάξουμε. Η συζήτηση είναι εξελισσόμενη. Αυτό είναι ένα από τα θέματα μάλιστα που θα συζητηθούν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 23-24 του Ιουνίου. Και νομίζω ότι τα κράτη-μέλη όχι μόνο θα έπρεπε να εγκρίνουν την πρόταση που έχει υποβληθεί για την ενίσχυση του Frontex, αλλά και να δώσουν στη διάθεση του Frontex περισσότερες δυνατότητες, αεροσκάφη, πλοία. Δεν μπορούμε αυτά να τα έχουμε από τον δικό μας προϋπολογισμό. Και γι' αυτό πιστεύω, πιστεύω ότι υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά θα πρέπει να γίνει συντονισμένα οι προσπάθειε ε, ξεκίνησαν από την Επιτροπή η κυρία Μάλστρομ συνεργάζεται σχετικά με τα κράτη-μέλη και ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στι 23 και 24 Ιουνίου θα επιβεβαιώσει την προσέγγιση αυτή. Ταυτόχρονα χρειάζεται βέβαια και η συνεργασία των τρίτων χωρών. Είχα επισκεφθεί την Τινησία πρόσφατα, μίλησα με τον Πρωθυπουργό. Μα υποσχέθηκαν οι η συνεργασία, συνεργάζονται Τώρα προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε κάποιες ε, ρεαλιστικές συμφωνίες για τις υποδομήσεις. Ευχαριστώ. Λείπουν αρκετοί ευρωβουλευτές λόγω του συναγερμού. Ο κύριος Φερχόφστατ θα θέσει το επόμενο ερώτημα. Βλέπω ότι κάποιοι από τους συναδέλφους είναι ακόμα στην άσκηση πυρασφάλειας. Ε, Uh, Συνάδελφοι, χθε ο επίτροπο κύριος Ρένα ανήγγειλε μια σειρά σημαντικών βημάτων στην Επιτροπή. Ένα μηχανισμό διάσωση, ζήτησε μάλλον αλλαγέ στο μηχανισμό διάσωσης, είπε ότι είναι αναγκαίο ο μηχανισμός αυτός να παράσχει πιστώσει ευέλικτε στα κράτη-μέλη, δυνατότητα να πάει στο δεύτερο πακέτο ο μηχανισμός και είπε ιδίω ότι τούτο μπορεί να γίνει με, ε, με swap εκπτώσεων σε, σε με bonds, με, με, με ομόλογα 3α, τριπλό α. Κάτι πολύ σημαντικό που επιτρέπει να αποκτούν τέτοια ομόλογα χώρες που είναι σε κίνδυνο. Επίσης είπε ότι θα εξετάσει το ενδεχο... η Επιτροπή θα ξεκινήσει να εξετάζει το ενδεχόμενο των ευρωομολόγων. Επιτέλους θα έλεγα εγώ. Η ερώτησή μου κύριε Πρόεδρε είναι μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι αυτή είναι η θέση της Επιτροπής. Δεύτερον πιέζει ο χρόνος Πρόεδρε θα προτείνετε τις αλλαγές αυτές για το, στο μηχανισμό διάσωσης στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε δύο εβδομάδες. Ευχαριστώ. Να επιβεβαιώσω ότι όλες οι ιδέες που παρουσίασε ο Επίτροπος κύριος Ρεν βεβαίως έχουν την πλήρη υποστήριξή μου. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν αυτά που είπε. Σε ό,τι αφορά τώρα τον μηχανισμό στήριξης αυτή τη στιγμή είναι υποδιαδικασία υλοποίηση. Θα συμφωνηθεί πολύ σύντομα ελπίζω. Ελπίζω λοιπόν ότι το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λάβει πολιτική απόφαση που θα επιβεβαιώνει τις αποφάσεις για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Και ξέρετε ποια είναι η θέση μας βεβαίως. Σε ό,τι αφορά τα ευρωομόλογα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και χρόνια και ένας προκάτοχό μου είχε προτείνει ευρωομόλογα. Η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη δεν δέχτηκαν την ιδέα αυτή. Τώρα, όταν εμφανίστηκε η κρίση στην Ελλάδα, προτείναμε μια αντίστοιχη ιδέα ε, του χρέου που δεν έγινε δεκτή από κάποια κράτη-μέλη τη ένωση Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει η διάθεση εξέταση διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. Η Επιτροπή προέτεινε μια σειρά εναλλακτικών. Η ιδέα των ευρωομολογών ήταν ελκυστική εφόσον βεβαίως τα κράτη-μέλη μπορούσαν να την υποστηρίξουν. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση για να σας πω την αλήθεια και πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στον μηχανισμό. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω πρόεδρε ότι τελείωσε η κρίση με την Ελλάδα και το ευρώ. Άρα πρέπει να βρεθούν επιπρόσθετα μέσα. Ένα από αυτά είναι αυτό που προτείνει ο Όλι Ρεν. Ένα swap από ε, επισφαλή χρέος κάποιων χωρών σε ένα μικρό πακέτο ευρωμολόγων τριπλού α. Και αυτό μπορεί να εκδοθεί από τον προσωρινό μηχανισμό, από τον μόνιμο μηχανισμό, από μια ευρωπαϊκή μελλοντική υπηρεσία. Ε, δεν έχει σημασία ποιος θα τα εκδώσει, αλλά το αντικείμενο και για πρώτη φορά αναγνώρισε όλη η και Επιτροπή ότι αυτό είναι μια λύση. Κύριε Φεχόφστατ, η Επιτροπή δρά συλλογικά, ω συλλογικό όργανο. Εσείς μπορείτε να συμφωνήσετε με αυτό που λέει ο κύριος Ρεν και να μην συμφωνείτε με μένα, αλλά τα ίδια πράγματα λέμε. Η Επιτροπή στην ετήσια έκθεση ανάπτυξης υποστήριζε την ιδέα μεγαλύτερης παρέμβασης της Ένωσης στις αγορές, κάτι που δεν δέχθηκαν δυστυχώς τα κράτη-μέλη. Αυτό που μπορώ να επιβεβαιώσω σε εσά είναι ότι πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση αυτή, προσπαθούμε να αυξήσουμε τις δυνατότητες ευέλικτης παρέμβασης στην αγορά, άρα ειλικρινώς πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να, δώσουμε έμφαση στον ευρωπαϊκό μηχανισμό και να δούμε το μέλλον των ευρωμολόγων αργότερα, εάν συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη. Ο κ. Σαχράντιλ. Θα μιλήσω τσέχικα, πρόεδρε. Pane předsedo Barroso, jak víte, moje skupina je složena... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική μου ομάδα αποτελείται ε, κυρίως από βουλευτές που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωζώνης. Από την άλλη εμείς δεν ευχόμεθα μία αποτυχία του ευρώ φυσικά. Οι οικονομίες μας είναι ιδιαίτερα αλληλοσυνδεδεμένες και μια τέτοια αποτυχία θα είναι κακή για όλους. Η, τα αισθήματα τα οποία έχουμε για τα τελευταία γεγονότα είναι ανάμεικτα. Από τη μία βλέπουμε αντιφατικές δηλώσεις από πλευρά του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμπεριφέρεται διαφορετικά, το Δέλτα Νιτάφ έχει μια διαφορετική λογική και έχω τελικά την αίσθηση ότι ε, τελικά υπάρχουν ορισμένες υποβόσκουσες πολιτικές αντιθέσεις και όχι οικονομικές απόψεις οι οποίες επικρατούν. σχετικά τώρα με την αναδιάρθρωση των χρεών των κρατών που έχουν προβλήματα. Ποια είναι η θέση σας. Προτιμάτε πάντα να υπάρχουν δανειοδοτήσεις όλο ένα πιο μεγάλες προς τις χώρες αυτές χωρίς ε, διαβλεπόμενο τέλος αυτών των διαδικασιών. Γιατί αναφέρομαι σε οικονομίες οι οποίες έχουν τρομακτικά προβλήματα είναι λίγο πριν από τον κρεμό ή μήπως έχετε αρχίσει να λογικεύεστε και έχετε αρχίσει να στρέφεστε και προς άλλες λύσεις. Ξεκινώντας κύριε Τσαχράντιλ, ε, ασχολούμεθα όχι μόνο με τη ζώνη του ευρώ αλλά και με ε, χώρες ε, εκτός της ζώνης ευρώ οι οποίες και αυτές κάποιες από αυτές τις χώρες είναι σε διαδικασίες βοήθειας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ. Υπάρχουν συζητήσεις οι οποίες συνεχίζονται ανάμεσα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να υπάρξει μια πλήρης απάντηση στο πρόβλημα. Συνεχίζονται οι συζητήσεις. Δεν υπάρχουν πάντα σαφέστατες συμφωνίες για τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει αυτή η απάντηση. Και γι' αυτό η διαδικασία είναι συνεχιζόμενη το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε είναι περίπλοκο, είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα και απαιτείται πολύ προσεκτική εργασία για να καταλήξουμε σε μια κάποια σύγκληση. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ επιφυλακτική όταν αναφέρεται στα θέματα αυτά γιατί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα τα θέματα αυτά. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα οποία είπαμε δεν είναι εναλλακτική λύση στις οδυνηρές διαδικασίες οικονομικής, δημοσιονομικής μάλλον εξυγίανσης, στις οποίες θα πρέπει να περάσουν τα κράτη-μέλη που έχουν τα προβλήματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Συμπρόεδρος κ. Σκονπεντήτ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Μπαρόσο, δεν καταλαβαίνει κανείς πολύ καλά την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα αυτά και μόλις γι' αυτά μιλήσατε. Καταρχά για το θέμα της αναδιάφρωσης. Κοιτάξτε, ε, ας μην κοροϊδευόμαστε. Κάποια στιγμή θα υπάρξει ε, μία αναδιάρθρωση του χρέους στην Ελλάδα σαν παράδειγμα για ένα απλό λόγο γιατί θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στην ελληνική κυβέρνηση συγκεκριμένη περίπτωση να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της και να αναδιαρθρώσει την ελληνική κοινωνία γιατί σήμερα στην Ελλάδα κανένας δεν εμπιστεύεται κανέναν και δεν εμπιστεύεται και την κυβέρνηση και αν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να δώσει μια προοπτική στον λαό της εκτός από τη λιτότητα τότε προφανώς δεν θα μπορέσει να ανακάμψει η οικονομία. Συνεπώς θα πρέπει στις σκέψεις τις οποίες κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε εμπιστοσύνη εκ νέου στον ελληνικό πληθυσμό στους Έλληνες πολίτες είναι η προϋπόθεση για να μπορέσουν τα μέτρα να έχουν κάποιο νόημα. Γιατί σήμερα με όλα αυτά τα μέτρα λιτότητας η κοινωνία δεν έχει ανάσα πλέον και γι' αυτό μπορεί να σημειωθεί μια πολύ μα πολύ επικίνδυνη άρνηση από πλευράς της. Δεύτερο θέμα, φοροδιαφυγή δεν μπορεί εν πάση περιπτώσει η Ευρώπη να βοηθήσει την Ελλάδα στον τομέα της φοροδιαφυγής. Έχετε τράπεζες στην Αυστρία, στο Λουξεμβούργο, στην Κύπρο βεβαίως και στην Ελβετία όπου υπάρχουν λογαριασμοί πολύ μεγάλοι Ελλήνων. Γιατί να μην παγώσουν αυτοί οι λογαριασμοί. Γιατί να μην τεθεί λίγο σε παρένθεση το πιστοτικό απόρριτο έτσι ώστε να μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει τη φοροδιαφυγή γιατί θυμίζω ότι οι Ευρωπαϊκέ τράπεζε, οι δικέ μα τράπεζε καλύπτουν τη φοροδιαφυγή. Δύο λεπτά μιλήσατε κύριε Πρόεδρε. Φταίει, φταίει η πυρκαγιά, φταίει η λέει ο κύριος Κονπεντήτ. Κύριε Κονπεντήτ, πράγματι υπάρχει θέμα φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Αν και δεν είναι αυτή η αιτία του διαφθορτικού προβλήματο που χαρακτηρίζει αυτή τη χώρα. Στη συγκεκριμένη φάση προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με το απόρριτο το τραπεζικό. Ξέρετε ότι όλες οι χώρες και η Ελβετία από το Μάρτιο του 2009 αποφάσισαν να εφαρμόσουν τα επίπεδα του ΩΣΑ έτσι ώστε καμία χώρα μέλη να μην μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες σε ένα άλλο κράτος μόνο και μόνο γιατί η πληροφορία αυτή κατέχεται και ελέγχεται από ένα πιστοτικό ίδρυμα. Η αρχή αυτή έχει συμπεριληφθεί και στην οδηγία για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 11 Μαρτίου του 2011 και θα τεθεί σε λειτουργία δυστυχώς μόνο την 1η Ιανουαρίου του 2003. Συνεπώς το θέμα του τραπεζικού απορρίτου έχει επιληθεί σε επίπεδο νομικό δεν μπορεί να είναι εμπόδιο σε ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών. Και γι' αυτό ακριβώς σήμερα, στα πλαίσια αυτής της δικατικής μορφής συνεργασίας, τα κράτη-μέλη να δώσουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται προς την Ελλάδα στον τομέα της πιθανής φοροδιαφυγής ή φορολογικής απάτης. Ο κύριος Μπίσκι. Α, όχι, συγγνώμη. Ε, κύριε Κονπεντή, δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο. Χρησιμοποίησατε όλο το χρόνο σας. Okay, we'll receive. Well, please. Ich kürze. Ναι, παρακαλώ. Θα είμαι εγώ πιο σύντομο, έτσι, συναδελφικά αφαιρόμενο. Κύριε Μπαρόζο, έχω μία σύντομη ερώτηση. Χαίρομαι που εξετάσετε το θέμα του διαδικτύου στην διασκέψη κορυφή ε, ε, του G8 έχει κανένας βέβαια ανησυχίες γιατί οι ισχυροί ασχολούνται με το διαδικτυό. Ξέρουμε πως ο ο τομέας. μπορεί να μας πείτε κάτι παραπάνω, ήταν μοναδική περίπτωση, θα ξανατεθεί στην ημερησία διάταξη. Κοιτάξτε, ήταν μια ιδέα του Πρόεδρου Σαρκοζή, θαυμάσια ιδέα μου φαίνεται, γιατί είναι παγκόσμιο επίπεδο του διαδικ... ε, φαινόμενο του διαδικτύου. Θέλουμε μια δυνατότητα ανοιχτού διαδικτύου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καμιά φορά όμως υπάρχουν καταχρήσεις στο διαδικτύο Εκμετάλλευση, παραδείγματο χάρη παιδιών. Εγκλήματα. Μέσω των ελευθεριών που δίνει το διαδίκτυο υπήρξαν λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει μεταξύ μερικών των μεγάλων δημιουργών πρωτοβουλειών στο πλαίσιο του ο, ο διαδικτύου κεφαλής του ο, FaceNet και άλλων. Ε, θέλησαμε λοιπόν να δούμε τι μπορεί ε, να γίνει για να προστατεύσουμε διατηρώντας όλες τις δυνατότητες καινοτομίας και θα είναι στο μέλλον ξανά το θέμα αυτό του διαδικτύου στην μέση εντάξει του G8. Στην πραγματική ερώτηση του κ. Πίσκελ. Κύριε Πρόεδρε, θα παραμείνω προσεκτικό για το θέμα αυτό και θέλω να σα ρωτήσω κατά πόσον προτίθεστε να μας, να, να ενημερώνετε για τις μελλοντικές επραγματεύσεις για το διαδίκτυο και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον μας. Μα δεν, δεν έγινε διαπραγμάτευση, είναι η απάντηση. Υπήρχε μια πολύ γενική ανταλλαγή απόψεων, ένα είδο brainstorming, αν μπορούμε να το πούμε, θύελα εγκεφάλων. Υπάρχουν οι μεγάλοι ενδιαφερόμενοι τη βιομηχανία ε, του διαδικτύου και με, με, με πολιτικούς σε μια μεγάλη διάσκεψη. Δεν ήταν διαπραγμάτευση. Εγώ το θεώρησα σαν διαπραγμάτευση. Εμείς ζητήσαμε από τους μεγάλους υπευθύνους της βιομηχανίας του διαδικτύου να μας πούνε πώς βλέπουν το μέλλον και εμείς μέσα στα πλαίσια του G8 επίσης παρουσιάσαμε δικέ δικές μας αποστάσεις, ε, συμπεράσματα, συμφέροντα κλπ. Χωρίς απορροφή. Ο κύριος Φάλιας έχει τον λόγο. Πρόεδρε, είχαμε μια σειρά ε, παντομιμικών ανταλλαγών. Κάποτε κάθε φορά σας έλεγα πάμε σε πτώχευση, μας λέγατε όχι δεν πάμε σε πτώχευση. Τώρα φτάνουμε στην τέταρτη που είχατε πει ότι δεν χρειαζόταν. Η ερώτηση που σας θέτω είναι πιο σοβαρή. Όχι αυτή που συνέβη στην Ελλάδα ή την Πορτογαλία ή την Ιρλανδία. Η πραγματική κρίση που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Την ακαιρεότητα της, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν μπορούμε δεν μπορείτε να συνεχίσετε να εξαγοράζετε τεράστιες ποσότητες του δικού σας επισφαλούς χρέους. Δέχεστε κύριε Μπαρόζο ότι η, η ακαιρεότητα και η οικονομική ακαιρεότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Όχι. Δεν το δέχομαι. Η Κεντρική Τράπεζα είναι εξαιρετικά αξιόπιστο θεσμικό όργανο με μεγάλη εξυπνάδα και φρονιμάδα λειτουργεί. Η ανεξαρτησία της είναι σεβαστή από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώ, του, της, ζώνη, της Ευρωζώνης. Υπάρχουν δυσκολίες στην Ευρωζώνη. Οι δυσκολίες αυτές δεν είναι μόνο της Ευρωζώνης, το είπα και προηγουμένω. Οι επικρίσεις είναι ιδεολογικού χαρακτήρα πάντα. Το πρόβλημα του χρέους δεν είναι αποκλειστικό της Ευρωζώνης. Κατά μέσο όρο το χρέος ε, των χωρών της Ευρωζώνης είναι χαμηλότερο από της Βρετανίας για παράδειγμα. Υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα εδώ, διότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτού του είδους την νομισματική ένωση χωρίς πιο ενοποιημένο θεσμικό πλαίσιο. Αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με ενιαία προσέγγιση και προσπαθούμε να δώσουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ. Χτες το Think Tank Open Europe έδωσε κάποια νούμερα. Η έκθεση της τράπεζας 190 δις ευρώ αποτελεί έκθεση στο, ευρωπαϊκό, στο ελληνικό κράτος και τις ελληνικές τράπεζες. Μία τόση, κατά 4,5% θα, ε, της ε, Ευρωζώνης θα οδηγήσει σε εξάλληψη απόλυτα αυτού του ε, ποσού. Με την σοβαρότητα κατάσταση με τη σοβαρότητα της κατάστασης του ευρώ αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι μπορείτε να απαντάτε έτσι όπως απαντάτε. Πρώτον, δεν λέω ψεύδι, ε, πάντα ήμασταν συνεπείς στις πληροφορίες που δίναμε για την κατάσταση. Για κάθε κατάσταση. Η κατάσταση είναι δύσκολη, το είπαμε εξ αρχής. Δεν λέμε ότι είναι μια ωραιότατη κατάσταση. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αξιοπιστία διότι στηρίζεται στην αποφασιστικότητα των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης να κάνουν ό,τι μπορούν για την δημοσιονομική σταθερότητα της ζώνης και για τη βιωσιμότητα και για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Λοιπόν, δεν έχω καμία αμφιβολία ούτε για την ικανότητά της να προασπίσει το τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και την δέσμευση των κρατών μελών της Ευρωζώνης να παράσχουν όλες τις εγγυήσεις που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να τηρήσει τον ρόλο ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας. Και πρέπει να σας πω ότι πέραν της δικής μας άλλες κεντρικές τράπεζες εκτός Ευρώπης βρίσκονται σε πολύ πιο δύσκολη και ευάλωτη κατάσταση από ότι είναι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είναι αξιόπιστη σεβαστή διεθνώς στην Ένωση. Η κυρία Σινκλέρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ένωση γίνεται ευρύτερη με την δημιουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και την αδυναμία να πετύχει συνένεση. Η αντίθεση της, Ευρώ, της Γερμανίας στην κατάσταση στην ε, Λιβύη το δείχνει. Μπορείτε να με εξηγήσετε πώς είναι δυνατό να υπάρξουν κοινέ πολιτικέ σε σημαντικού τομεί διεθνών σχέσεων και ασφάλεια χωρί τη συνένεση. Εκτό εάν απαρνηθούμε τα δημοκρατικά δικαιώματα των κρατών ελών να ε, ε, ομονομερό να εφαρμόζουν τι δικέ του προσδοκίε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Είμαστε μια ένωση 27 δημοκρατικών χωρών και στα πλαίσια της ΚΕΠΑ, της κοινή εξωτερικής πολιτικής, και πολιτικής ασφάλειας έχουμε συμφωνήσει ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ε, ομοφόνος. Εάν δεν υπάρχει ομοφωνία τότε δεν έχουμε την δυνατότητα να επιβάλλουμε η αδίποτε απόφαση στα υπόλοιπα κράτη. Συνεπώς σεβόμεθα πλήρως την δημοκρατική φύση της Ένωσης και τις σχέσεις μας με τα κράτη-μέλη είναι προς όφελός μας και προς όφελος των πολιτών της Ένωσης τα κράτη-μέλη να δράσουν από κοινού τις εξωτερικές υποθέσεις της Ένωσης. Είναι προφανές, γιατί ακόμα και οι μεγαλύτερες χώρες δεν έχουν, αν θέλετε, την μεγαλύτερη δυνατότητα μόχλευσης και επιρροής χωρών όπως η ΙΠΑ και η Κίνα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού μπορεί να επηρεάσει. Και γι' αυτό ελπίζω η διαδικασία να οδηγήσει σε μεγαλύτερη σύγκληση και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Ευχαριστώ συμπληρωματική ερώτηση της κυρίας Σίνκλα. Κοιτάξτε, εγώ μίλησα για τα πανευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί ο Ευρωπαίος φορολογούμενος να χρηματοδοτεί αυτού του είδους τα κόμματα και τι χρησιμότητα έχουν τα κόμματα αυτά για τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μια ερώτηση για την κάθε άστον ξέρω ότι δεν συμμετέχει πολύ στις συναντήσεις των επιτρόπων. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Ξέρετε ότι είναι αναγνωρισμένα σαν σημαντικές οντότητες από τη συνθήκη η οποία επικυρώθηκε ομόφωνα από τα κράτη-μέλη. Συνεπώς υπάρχει λόγος υποστήριξης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, διότι πράγματι είναι ευρωπαϊκές οντότητες που αναγνωρίζονται από τη συνθήκη. Για την κάθε άστον Ξέρετε ότι δεν είναι μόνο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά είναι και ότι εκπρόσωπο στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Έχει μια πολύ δύσκολη δουλειά, εκφράζει και αντιπροσωπεύει την Ένωση στο εξωτερικό και έχει πολύ περισσότερες αποστολές από όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθεί να συμμετέχει σε όλα τις συναντήσεις των Επιτρόπων, δεν τα καταφέρνει βέβαια, αλλά να θυμίσω ότι η κυρία Αστων όπως και όλοι οι Επίτροποι δεν εκπροσωπούν τις χώρες τους, αλλά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακριβώς εμείς δίδουμε όρκο όταν αναλαμβάνουμε την υπηρεσία μας και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδράζεται ακριβώς στην προσπάθεια του να είμαστε ανεξάρτητοι και ε, το Ηνωμένο Βασίλειο σαν παράδειγμα αντιπροσωπεύεται πάρα πολύ καλά στο Συμβούλιο και ε, στη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σούλτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Παρακαλώ, συγχωρήστε την καθυστέρησή μου. Έπρεπε κάτι να ολοκληρώσω. Κύριε Μπαρόζο, λόγω τη σοβαρή κατάσταση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Το 2008 είχαμε μία τραπεζική κρίση η οποία οδήγησε το 2009 σε μια βαθιά οικονομική κρίση της οικονομίας. Η ανάληψη του κόστους ε, από τα κράτη οδήγησε το 2010 σε μια βαθιά κρίση των δημοσίων οικονομικών που οδήγησε σε μια περικοπή, σε ένα όριο περικοπών που εν μέρει το ζητήσαμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξ αυτού σε ορισμένε χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δημιουργήθηκαν διαρματικέ καθιστάσει. Υπάρχει κίνδυνο το 2011 και 2012 μετά από την κρίση των τραπεζών, της οικονομίας και των ε, δημοσίων οικονομικών θα υπάρξει μια κρίση κοινωνική. Σας ρωτώ λοιπόν, προτίθεται η Κομισιόν να συζητήσει το θέμα από κοινού με εμάς ε, Πώς θα μπορέσουμε δηλαδή η ανεπαρκής χρηματοδότηση των κοινωνικών αναγκών στα κράτη-μέλη, ιδίω εκείνες χώρε που πλήττονται περισσότερο από τι ε, δημοσιομικές κρίσει, θα μας βοηθήσετε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη χρηματοδότηση αυτών των συστημάτων. Και επίσης να το θέμα των ευρωομολόγων για να αποκτήσουμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε για να επενδύσουμε στις ε, οικονομίες μας, για να μπορέσουμε να δώσουμε δυνατόν να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης ε, στις ε, χώρες που έχουν επιλογή περισσότερο. Τον Ιούλιο η Κομισιόν υιοθέτησε μία ανακοίνωση για κάθε χώρα και μία ανακοίνωση η πιο γενική που καλύπτει ακριβώς αυτό το σημείο που αναφέρατε. Είναι για μα αυτό πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξέρουμε ότι η λιτότητα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να μειωθεί το έλλειμμα και το χρέος είναι περίοδοι πάρα πολύ δύσκολη. Και θεωρούμε ότι κάθε ένα ευρώ που δαπανάτε αυτή τη στιγμή για την εξυπηρώτηση του χρέους είναι ένα ευρώ που λείπει από τα ε, νοσοκομεία, από τη δημόσια ε, τα δημόσια νοσοκομεία από την κοινωνική ασφάλιση. Και γι' αυτό πρέπει να γίνουν σημαντικότατες ε, προσπάθειες για να διατηρηθεί μια ισορροπία και ταυτόχρονα να προστατευτούν βέβαια οι πιο ευάλωτες ε, ομάδες ε, των πληθυσμών. Και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε περισσότεροι να εργαστούν στην αγορά εργασίας πώς θα δώσουμε αυτή την κοινωνική διάσταση σε όλη την οικονομία για να δούμε πώς μπορούμε να εγγυηθούμε αυτούς τους στόχους που συμμεριζόμαστε νομίζω. Ευχαριστώ. Διαδικασία Κατσουδιάλη ο Πρόεδρος. Λυπούμε. Μη ένα λεπτό και μετά δύο δευτερόλεπτα την ερώτησή σας. Δεν έχουμε πια χρόνο. Όπως είπα και στον κύριο Κονμπένιτ και στον κύριο Σαγράτιο. Δεν τους έδειξα τη δυνατότητα για την πραγματική ερώτηση. Λυπούμε. Κάτσε δε Εκτός μου κύριο Σούρτ. Well, but uh, Έχουμε κανόνες κύριε Πρόεδρε, τι να κάνουμε. Λυπούμε. Λυπούμε πραγματικά. Κάτσε διάει. Σύνοδος της ομάδος των 8, του G8. Ο κύριος Μάρκος Κούρια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν ήθελα να μιλήσω για τους G8. Να θέσω ένα ερώτημα για θέματα πολιτισμού στον κύριο Μπαρόζο. Έχουμε στην Ένωση πολλά προγράμματα που ενθαρρύνουν νέους και όχι μόνο να συναντιούνται ούτως ώστε να μετατρέψουμε την Ένωση σε πραγματική Ένωση. Comenius, UNAction, και κλπ. που για πολλούς νέους επαγγελματίες ήταν η πραγματική συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διακόπτε το μιλητής. Κοιτάξτε, το θέμα μας είναι η ομάδα των 8. Παρακαλώ συνεχίστε. Λάθος ανακοινώσεων τέλο πάντων. Έλεγα, κατά την άποψη της Επιτροπής, τι μέλλον έχουν τα προγράμματα αυτά που λήγουν και κανονικά θα έπρεπε να, έχουμε ήδη εξετάσει στην Επιτροπή Πολιτισμού. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να αναπτύξει μετά το 2014 την επόμενη περίοδο προγραμματισμού τα ζητήματα αυτά, γιατί πιστεύω ότι αυτά ενδιαφέρουν πολλούς νέους και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή ενδιαφέρεται προφανώς για την πρόθεση της πολιτισμικής διάστασης στην Ευρώπη και εγώ προσωπικά το θέλω. Ήδη συνάντησα κάποιους από τους βασικούς δρόντες στον τομέα. Αυτό που θα κάνουμε είναι να υποβάλουμε στο τέλος του μήνα προτάσεις ούτως ώστε για τις δημοσιονομικές προσωπικές αλλά σε όλους τους κλάδους με συγκεκριμένες σημαντικές προτάσεις. Θέλουμε να εξορθολογήσουμε τα εργαλεία αλλά εξασφαλίζοντας τις φιλοδοξίες μας, ιδίως για τα προγράμματα που αναφέρατε και που είναι εμβληματικού χαρακτήρα, πολύ σημαντικά για τη δημιουργία μιας Ευρώπης πολιτών, μιας Ευρώπης που θέλει να διατηρήσει τις ευρωπαϊκές αξίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Λάτφολτ. Θα μείνω στο ίδιο θέμα, Πρόεδρε. Χτες η Επιτροπή υιοθέτησε ένα μεγάλο πακέτο μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς που κοστίζει 120 δις ευρώ το χρόνο, περίπου όσο και ο προπολογισμό της Ένωσης. Ωστόσο, πολλά κράτη-μέλη, οκτώ κράτη-μέλη παίρνουν χαμηλό βαθμό στον δείκτη της διεθνούς διαφάνειας. Για να Μήπως θα έπρεπε λοιπόν στη σύνοδο των 8, του G8 να τεθεί και το θέμα της διαφθοράς. Η μόνη όμως μνήμα που είδα στις ε, αναφορές ήταν για τις αναπτυσσόμενες χώρες, όχι για το πώς πρέπει να δείξουν οι πλούσιες χώρες την πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στο σπίτι τους. Μήπως ήταν μια ευκαιρία χαμένη για να συζητηθεί το θέμα της διαφθοράς και της δωροδοκίας των G8, ιδίω όταν η Ρωσία, ένα μέλος, είναι 148, νούμερο 150 κάτι, στον δίκτυο αυτό. Ευχαριστώ. Το θέμα της διαφθοράς δεν τέθηκε στη συνάντηση με τους Αφρικανούς ηγέντες, αλλά θα είναι στην ομάδα, στην ημερήσια διάταξη του Νοέμβριο του G20. Ξέρετε, όταν έχουμε διαφθορά, κάποιος διαφθείρεται, αλλά για κάποιος διαφθείρει. Άρα και η ομάδα των 8 εξετάζεται όταν συζητούμε το θέμα αυτό. Και έγινε. Και έχω και καλά νέα να σας πω, διότι είπε ότι η Επιτροπή θα υποβάλει πρωτοβουλίες στον τομέα της διαφάνειας για τις πρώτες ύλε. Καλό παράδειγμα αντιμετώπισης ε, προβλημάτων όπου σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαφάνεια οδηγεί ευκολότερα κάποια καθεστώτα να χρησιμοποιούν χωρίς μεγάλο έλεγχο εθνικούς πόρους προς του αναπτυγμένου κόσμου στις πολλές περιπτώσεις. Άρα από αυτή την οπτική γωνία συζητήθηκε στο G8. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαντάλεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση, αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την οποία χαρακτηρίσατε ανεξάρτητη. Αλλά δεν είναι πλήρως ανεξάρτητη και δεν στάθηκε ανεξάρτητη στην κρίση την ελληνική σαν παράδειγμα λειτουργήσε σαν εμπορική τράπεζα, αγόρασε δισεκατομμύρια ομόλογα και τώρα είναι εναντίον των απαραίτητων αναδιαρθρώσεων, της απαραίτητης μάλλον αναδιαρθρώσεως της, Ευρωπα... της ε, ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα με αυτόν τον ρόλο, τον διπρόσωπο κατά κάποιο τρόπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση με την ε, χρειαζόμενη ελληνική αναδιάρθρωση είναι ανεξάρτητη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ανεξαρτησία αυτή αναγνωρίζεται από τις συνθήκες. Μετά από 7 χρόνια εμπειρία στη συγκεκριμένη θέση, έχω έρθει πολύ συχνά σε επαφή με την Κεντρική Τράπεζα και τον πρόεδρο φυσικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δεν χρειάζεται την ε, βοήθειά μας για να επιβεβαιώσουν την ανεξαρτησία τους σχετικά με την αναδιάφρωση του χρέους. Όπως ξέρετε υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και επιλογές στα πλαίσια των αναλυτών. Εμείς ε, λαμβάνουμε υπόψη μας όλα όσα λέγονται στις συζητήσεις, αλλά η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Θεωρούμε ότι δεν είναι εναλλακτική λύση η αναδιάρθρωση στις προσπάθειες τις οποίες θα πρέπει να κάνουν τα μέλη για την δημοσιονομική τους εξυγίανση. Αυτή ήταν η αρχική μας θέση, συνεκτική θέση και θα εμείνουμε σε αυτή. Η κυρία Φιγουερέδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην τελευταία συνάντηση της ομάδας των 8 θα ήθελα να μάθω κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εάν για μια ακόμη φορά τέθηκε σε αναβολή, δεν έγινε η συζήτηση εν περιπτώσει το θέμα της φορολογίας της κίνησης των κεφαλαίων, των υπεραξιών και των φορολογικών παραδείσων και αν ασχοληθήκατε με το θέμα των υπηρεσιών αξιολόγησης οι οποίες αυτή τη στιγμή ε, λειτουργούν χωρίς καμία διαφάνεια και των οποίων ε, οι εργασίες γενικά δεν θεωρούνται αξιόπιστες. Όλα αυτά, ξέρετε, συνδέονται με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ολλανδία και η Ελλάδα. Εμείς στην ουσία το μόνο που κάνουμε είναι να επιβάλλουμε στους εργαζομένους των χωρών αυτών κάποιες διαδικασίες και κάποια μέσα τα οποία δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να χειροτερεύουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Καταστάσεις επιβαλόμενες εκ των άνω οι οποίες οδηγούν σε περαιτέρω οικονομική ύφεση και οι οποίες μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οδηγούν στην ανεργία, στην φτώχεια και στην ανισότητα. Πράγματα εντελώς αντίθετα και αντιφατικά σε σχέση με αυτά τα οποία στηρίζει η συνθήκη. Κυρία Φιγηρέδο. Καταρχάς, σχετικά με τα θέματα της ρυθμίσεως των χρηματαγορών και στην ομάδα των 8 και στην ομάδα των 20 έχουμε αρχίσει να συζητάμε ότι θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε γύρω από την υπόθεση αυτή. Εγώ ο ίδιος στα πλαίσια της ομάδας των 8 ξεκίνησα μια συζήτηση. Μια συζήτηση για την πιθανή φορολόγηση ε, ε, ε, των, συναλλαγών σε τομέα χρηματοοικονομικό. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές απόψεις υπέρ της δημιουργίας ενός τέτοιου φόρου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ορισμένες προτάσεις ταχύτατα. Γύρω από τις γενικότερες ερωτήσεις τις οποίες θέσατε, προφανώς και συζητήσαμε την κατάσταση σε ορισμένες χώρες της ζώνης ευρώ αλλά από την άλλη θεωρούμε ότι εφόσον υπάρξει μια ουσιαστική δημοσιονομική εξυγίανση, εφόσον δεν υπάρξει, τότε δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Στην συνάντηση της ομάδας 8 συζητήθηκε το θέμα της πολιτικής γειτονίας στη Μεσόγειο. Εσείς ε, δεσμεύσατε ε, ένα σημαντικό ποσό για τις πολιτικές 1,24 ε, δισεκατομμύρια για την πολιτική γειτονία που θα μπορούσα να πείτε ότι είναι μόνο για τον όχο. Ξέρουμε ότι στην αρχική πρόταση της Επιτροπής 150 εκατομμύρια πήγαιναν για την Ανατολή και τα υπόλοιπα για τον Νότο. Αυτό έχετε σε αντίφαση με την αρχή της συμμετρίας και της ε, ισότιμης αντιμετώπισης όλων των γειτόνων. Για, πώς το εξηγείτε αυτό γιατί δώστε τόσα πολλά για την πολιτική προς τον Νότο με τα πολύ λίγα χρήματα που είχατε στο συγκεκριμένο τομέα. Να σας πω ειλικρινώς, κύριε Βόλσκι, κατανοώ τις ανησυχίες που έχετε σε ό,τι αφορά την πολιτική γειτονία. Το πιο σημαντικό θέμα ωστόσο δεν είναι να φέρνουμε σε ανταγωνισμό την Ανατολή και τον Νότο, αλλά χρειαζόμαστε και τους δύο. Είναι σημαντικό να βοηθήσουμε αυτούς που θέλουν βοήθεια και με αποτελεσματικό τρόπο. Η προσέγγιση που υιοθετήσαμε στην αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας είναι σαφής. Δεν δίνουμε πόρους ανάλογα με το αν κάποια χώρα είναι στην Ανατολή ή στον Νότο, αλλά με, το, με την πρόοδο που έχει πετύχει κάποια χώρα. More for more, περισσότερο για περισσότερο. Όσο κάνεις περισσότερο, τόσο περισσότερο αξίζεις να λάβεις. Δεν έχουμε λοιπόν πακέτο προκατασκευασμένο για την Α ή τη Β χώρα. Κάθε χώρα πρέπει να δείξει ότι αξίζει τα κονδύλια που δίνουμε για αυτήν. Και στο πλαίσιο αυτό τηρούμε και τις δεσμεύσεις μας και προς τους γείτονες της Ανατολικής Ευρώπης και τους γείτονες στην, ε, στο Νότο. Κύριε Ντεσσαρνέζ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ερώτησή μας σχετίζεται με την προηγούμενη ερώτηση και την απάντησή σας. Απαντήστε στην ενίσχυση που δίνεται στις ε, αναπτυσσόμενες ε, αραβικές δημοκρατίες. μεταξύ άλλων περίπου 15 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και αναφερθήκατε στους διάφορους όρους και αυτή είναι η ερώτησή μου. Αυτή η βοήθεια εξ, εξαρτάται από κάποιους όρους, δηλαδή ελεύθερες εκλογές, καταπολέμηση της διαφθοράς, ανεξαρτησία της ε, δικαιοσύνης, ε, μεταρρύθμιση αστυνομίας ε, και του στρατού και όλα αυτά τα γνωρίζετε. Εγώ θέλω να ξέρω Ποιος θα αξιολογήσει για όλες αυτές τις αναδυόμενες αραβικές δημοκρατίες το σεβασμό των κριτηρίων. Θα εμπλακεί πλήρως το κοινοβούλιο μας για την αξιολόγηση αυτών των όρων ή θα υπάρχει μία ή θα είναι αρμοδιότητα στο Συμβούλιο. Απάντηση του κ. Περόζο. Η ερώτησή μας είναι ότι θα είναι επικεφαλής της άσκησης αυτής η Κομισιόν και είμαι πολύ περήφανος που η Κομισιόν με την ύπατη εκπρόσωπο υπέβαλε ακριβώς αυτή την, την απάντησή μας. Η τελική σχέση με τις χώρες αυτές της Μεσογείου. Και σήμερα στο Συμβούλιο αναγνωρίζεται ότι είναι καλό η Κομισιόν να βρίσκεται επικεφαλή της άσκησης αυτής. Και βέβαια η Κομισιόν είναι υπόλογη προς το Κοινοβούλιο. Όλες οι προσπάθειες δηλαδή του Κοινοβουλίου θα μπορούν να πληστούν πλήρες, πλήρως υπόψη. Έχουμε εδώ μια προσπάθεια στρατηγικής σημασίας, όχι μόνο για τι χώρες αυτές, αλλά για όλο τον κόσμο, είναι ανάπτυξη του μουσουλμανικού κόσμου και για μας στην Ευρώπη. Οι δικέ μας ε, κοινωνίε ε, θέλουν να υποστηρίξουν την μετάβαση αυτή στους γείτονές μας, παρά που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορώ παρά να χαιρετήσω το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου. Ο κ. Τινόκολας Αλαβράκος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, επ' ευκαιρία της Συνόδου των G8 διάβασα οικονομικά στοιχεία του 2009 σύμφωνα με τα οποία το παγκόσμιο ΑΕΠ ήταν 58 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το χρηματοοικονομικό χρήμα ανερχόταν στα 615 τρισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, στο θέμα νομισματική πολιτική που σας απασχόλησε, επιβεβαιώθηκε ότι οι ΗΠΑ εκδίδουν νέο χρήμα, νέα δολάρια, ενώ η Ένωσή μας δεν εκδίδει νέο νόμισμα. Ε, οι οικονομολόγοι διαφωνούμε σε πολλά πράγματα όμως δύο πράγματα μας έχει διδάξει η ιστορία ότι τον πτωχευμένο δεν τον σώζεις δίνοντάς του ακριβά δάνεια και το δεύτερο τη βαριά λιτότητα δεν μπορεί ποτέ να την μειώσει το έλλειμμα μιας μακροοικονομίας που βρίσκεται σε ύφεση και η οποία δεν μπορεί να υποτιμήσει το νόμισμά της. Το, ευρωνόμισμα, το, ευρωομόλογο κύριε πρόεδρε καθίσταται επιτακτικό. το βλέπετε σαν μέσον αντισταθμίσεως της ραγδαίας εκδόσεως νέου νομίσματος από τη ΣΥΠΑ. Ευχαριστώ. Δεν είμαι βέβαιος ότι όλες οι ερωτήσεις σχετίζονται αυστηρά με τη συνάντηση της ομάδας των οκτώ. Ίσως κάποιες παρατηρήσεις, κάποια στοιχεία να είναι παρόμοια. Ο κύριος Μπαρόζο, όντως, στο πρώτο τμήμα της συζήτησης θα έπρεπε να τεθεί αυτό το ερώτημα. Να απαντήσω ωστόσο στον κύριο βουλευτή η θέση της Επιτροπής τα τελευταία χρόνια ήταν ανοιχτή, θετική στην ιδέα των ευρωμολόγων. Από ένα, ένας προκάτοχός μου ήταν αυτός που πρώτος πρότεινε ευρωμόλογα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπήρχε συμφωνία από πλευράς κρατών ελών. Τι συμφώνησαν τα κράτη μέλη τώρα, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας που θα γίνει ενδεχομένως ο πρώτος χρηματοοικονομικός οργανισμός στον κόσμο σε ό,τι αφορά την χρηματοοικονομική δύναμή του. Και εκεί θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Ταυτόχρονα είμαστε ανοιχτοί στο να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο βεβαίως πολλές εναλλακτικέ δυνατότητες για το ενδεχόμενο ευρωομολόγων εφόσον βεβαίως υπό τον όρο μάλλον ότι υπάρχει βούληση των κρατών μελών να εξετάσουν τη δυνατότητα αυτή που είναι πολύ σημαντικό και αποφασιστικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ για την απάντηση στην ερώτηση που ήταν προβληματικά συνδεδεμένη με το θέμα μας. Ο κ. Μπρόνς, ένα λεπτό. Η τελευταία συνάντηση κορυφής υποτίθεται ότι θα έρθουν 40 δι στην την Ασία και την Αίγυπτο για να ανατρέψουν τις δικτατορίες και για να βοηθήσουν την δημοκρατία. Η ομάδα των 8 είπε ότι θα βοηθήσει τις χώρες που θα προχωρήσουν όχι μόνο στη δημοκρατία αλλά και την οικονομία της αγοράς. Θέλουν αυτές τις χώρες, λέει η ανακοίνωση του 8, να μπορέσουν να δρέπουν τους καρπούς της παγκασμιοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείε μας θέλουν να πάνε εκεί, να βγάλουν χρήματα και να τα πάρουν πάλι πίσω. Δεν ξέρω ακριβώς ε, πώς θα πετύχετε τους στόχους αυτούς, οι οποίοι είναι σωστοί βέβαια σε μια πρώτη φάση. Το θέμα είναι να πούμε στις χώρες αυτές τι πολιτικές θα πρέπει να ακολουθήσουμε και τι πολιτικές ε, θα πρέπει να απορρίψουν. Βέβαια δεν έχουμε εμείς το δικαίωμα να δίνουμε μαθήματα προς τις χώρες αυτές. Θα πρέπει ίσως να εκφράζετε τις ε, ερωτήσεις σας λίγο πιο αργά γιατί μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στην απόδοσή τους. Κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με την προοπτική την οποία ακολούθησε η ομάδα των 8. Νομίζω ότι είναι κοινό συμφέρον όλων μας να έχουμε όχι μόνο ανοιχτές κοινωνίες αλλά και ανοιχτές οικονομίες στην Αίγυπτο και την Ισία. Οι χώρες αυτές είναι οι γείτονές μας και νομίζω ότι ο καλότερος τρόπος είναι να τις βοηθήσουμε μέσω του εμπορίου. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις οικονομικές τους ανάγκες εφόσον παραμείνουν οι οικονομίες αυτές κλειστές. Στις χώρες του Μαγκρέμπου όπως γνωρίζετε ε, το εμπόριο μεταξύ τους των χωρών του Μαγκρέμπ είναι ασήμαντο. Ε, τους ζητάμε να ανοίξουν τις αγορές τους σε εμάς, αλλά δεν εμπορεύονται μεταξύ τους. Λοιπόν, θα σας το στηρίξουμε. Αλλά θα πρέπει και εσείς να ανοίξετε τις οικονομίες σας, να προχωρήσετε σε μια ολοκλήρωση των οικονομιών σας και η πρόοδος των χωρών αυτών συνδέεται άμεσα με την δυνατότητά τους να ενσωματηθούν στην παγκόσμια οικονομία. Κοιτάξτε την Νοτιοανατολική Ασία. Ακόμα και χώρες που δεν είναι δημοκρατικές, λόγω του ότι άνοιξαν τις οικονομίες τους, μπόρεσαν να ενταχθούν στην παγκοσμιοποίηση και να κερδίσουν από αυτή. Ο συνάδελφο Γκαμπριέλη Αλμπερτίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τελική δήλωση της συνάντησης κορυφής της ομάδας των οκτώ σχετικά με τη Μέση Ανατολή επιβεβαίει ότι οι διαπραγματεύσεις είναι ο μοναδικός δρόμος για μια σφαιρική λύση διαρκή του Μεσονατολικού το Ισραήλ και το Παλαιστινιακό Κράτο θα πρέπει να σεβαστούν τι υπάρχουσε συμφωνίε συνεργασία και να απέχουν από μονομερει ενέργειε, οι οποίε θα διακόψουν και θα διαρρήξουν την πορεία προ την πρόοδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σημαντικό συνομιλητή τη ομάδα των 8 υποστηρίζει άραγε αυτή την δήλωση. Το μεταφέρατε στην Παλαιστινιακή πλευρά η οποία θέλει το Σεπτέμβριο να προχωρήσει μονομερό κατά τη διάρκεια των Ηνωμένων Εθνών σε συγκεκριμένο διάβημα. Ευχαριστώ. για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. 30 χρόνια θυμάμαι σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις το θέμα ετίθετο. Και ζητούσαμε και τις δύο πλευρές να ξεκινήσουν ουσιαστικό διάλογο για να υπάρξει αποτελεσματική έκβαση. Όλοι επενέσαμε τη νέα προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση του ζητήματος ως ε, βασική θεμελιώδου αλλαγή, Ωστόσο υπήρχαν αντιδράσει στι λεπτομέρειε λεπτομέρειες του νέου, της νέας και μεταξύ των οκτώ στο θέμα της συνεργασίας Χαμάς-PLO και το θέμα της επιστοφής στα πρώτα 67 σύνορα. Επίσης υπήρχαν κάποιες ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο της πρόσφατης προσπάθειας ε, του, του, των Παλαιστινίων να ζητήσουν ε, την αναγνώριση του κράτους στην επόμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ελπίζω η Ευρώπη να έχει, αυτό που να σας πω είναι, η Ευρώπη να έχει κοινή θέση στο ζήτημα αυτό. Αυτό συζητούμε και με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαλίκα Μπενά Ατού. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Μπαρόζο. Οι χώρε τη ομάδα 8 αποφάσισαν να δώσουν 40 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ισία και το Αίγυπτο όπω αναφέρθηκε ήδη. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ζητήσει μεγαλύτερη διαφάνεια και ανιχνευσιμότητα των ποσών αυτών, καθώς και μια καλύτερη διακυβέρνηση της βοήθειας αυτής, με έμφαση σε τέσσερα βασικά σημεία. Ένα, την εγγύηση του δημοκρατικού χαρακτήρα και την απόλυτη διαφάνεια στην ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Δύο, να διασφαλίσει το, σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και να αυξήσει τον ρόλο και την ικανότητα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολισών και να οργανώσουν μια μεταρρύθμιση του συστήματος ρύθμισης της βοηθείας με μεγαλύτερη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Μπαρόζο, η Ένωση πρέπει να εγγυηθεί την καλή υποδοχή και λήψη των ενισχύσεων αυτών από τους τοπικούς πληθυσμούς. Τι συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Κυρία Βουλευτά, είπατε αυτά που σκέφτομαι ακριβώς. Θα συμφωνούσα, απόλυτα συμφωνώ μαζί σας. Θα υλοποιήσουμε αυτά που μας λέτε. Με πολλά μέσα για να επαληθεύσουμε κατά πόσον οι δεσμεύσει των χωρών εταίρων εφαρμόζονται ουσιαστικά. Και όχι μόνο η Επιτροπή με τις υπηρεσίες της, αλλά και η ύπατη εκπρόσωπος θα επαγρυπνεί γι' αυτό. Θα υπάρξει ειδικό εισηγητή για την περιοχή αυτή από την ύπατη εκπρόσωπο που θα παρακολουθήσει την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Πιστεύουμε ότι στο, διά, πλαίσιο του διαλόγου αυτού μπορούμε να βοηθήσουμε τι χώρε αυτέ ενισχύοντα την συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών. Πρόσφατα είχα πάει στην Τινησία είδα εκπροσώπου τη κυβέρνηση και των πρωτών τη Δημοκρατία, αλλά και εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών, γυναικείε οργανώσει, συνδικάτα και είδα πόσο θεωρούν σημαντική την εμπλοκή μας όχι μόνο κυβερνητικά αλλά και μέσω της κοινωνίας των πολιτών. Το είπα και στην κυρία Τεσσαρνές. Πιστεύω ότι η δουλειά του Κοινοβουλίου θα βοηθήσει πάρα πολύ στις σχέσεις με τα κόμματα, τα κοινοβούλια και τον κόσμο σε αυτές τις νέες δημοκρατίες. Ο κύριος Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, στην πρόσφατη συνάντηση στο G8 συζητήσατε για την παγκόσμια οικονομία και συμφωνήσατε στο ότι επικεντρώνονται οι προσπάθειες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, την ανάρτηση των οικονομιών, την αντιμετώπιση της ανεργίας. Και όλα αυτά γίνονται προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Όμως, ε, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι αν δούμε το παράδειγμα της Ελλάδας, πρόσφατα δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βγαίνουν στις πλατείες και τους δρόμους γύρω γύρω από την ελληνική βουλή αυθόρμητα χωρίς καθοδήγηση αλλά με αγανάκτηση αναζητώντας αξιοπρέπεια και προοπτική και πρέπει κύριε πρόεδρε να συμφωνήσετε ότι καμία πολιτική δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική εάν δεν έχει τη στήριξη ή έστω την ανοχή της κοινωνίας. αυτή η πολιτική στην ελλάδα ουσιαστικά περιορίζεται σε ένα δίλημα μεταξύ εξαντλητικής λιτότητας ή χρεοκοπίας. σας ανησυχούν αυτές οι κοινωνικές εξελίξεις; είναι ένα μείζον πολιτικό θέμα. και τι θα έχετε να πείτε και τι μήνυμα θα έχετε να στείλετε σε αυτούς τους ανθρώπους που με μεγάλη αξιοπρέπεια με ειρηνικό τρόπο διεκδικούν μια προοπτική και, ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους, τις οικογένειες και τα παιδιά τους. Ευχαριστώ πολύ. Thank Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου με τον ελληνικό λαό. Αναγνωρίζω τις δυσκολίες τις οποίες βιώνει η χώρα του σήμερα. Πιστεύω παράλληλα ότι η ευθύνη των πολιτικών ηγητών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, είναι να δείξουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν το σωστό οι κόρε τους. Χωρίς την δημοσιονομική εξυγίανση και μεταρρυθμίσεις η Ελλάδα δεν θα βγει από αυτή την κρίση. Συνεπώς η πραγματικότητα είναι ότι κάποια οδυνηρά μέτρα είναι αναπόφευκτα στην Ελλάδα. Και οποιοδήποτε πιστεύει το αντίθετο και πρεσβεύει το αντίθετο ψεύδεται προς τον ελληνικό λαό. Το, η έκκλησή μου λοιπόν προς τους Έλληνες ηγέτες είναι να εξηγήσουν ακριβώς αυτό προς το λαό τους, να τους δείξουν τις δύσκολες επιλογές τις οποίες θα πρέπει να προβούν. Εγώ ήμουνα στην συνάντηση του Συμβουλίου που οδήγησε uh, στη μείωση του επιτοκίου των δανείων που δόθηκαν προς την Ελλάδα, αλλά από την άλλη ε, θα πρέπει και η Ελλάδα να κάνει τη δική της προσπάθεια μια ε, χώρα δεν μπορεί να ζήσει ε, για πάντα σε τόσο υψηλά επίπεδα χρέους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν φυσικά και η κυβέρνηση της Ελλάδας και η αντιπολίτευση της Ελλάδας και όλοι εμείς στην Ευρώπη. Τελευταία ερώτηση Μπάφτον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Μπαρόζο, χαίρο που θέσατε στην ομάδα των, το, το θέμα των προβλημάτων της Ευρωζώνης. Είναι κρίση, το ξέρουμε όλοι όπως και ο προηγούμενος ομιλητής ανέφερε ωστόσο, πολλά κράτη-μέλη είχαμε διαδηλώσει στη Μαδρίτη την περασμένη εβδομάδα, στη Λισαβόνα διαδήλωναν. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Μήπως κύριε Μπαρόζο ήρθε η ώρα να σηκωθείτε. Είπατε προηγουμένω ότι δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Να σηκωθείτε λοιπόν και να πείτε την αλήθεια ότι θα πρέπει να επιτραπεί στις χώρες αυτές να φύγουν από την Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Σέβομαι τα δημοκρατικά κράτη της Ένωσης. Εγώ λοιπόν δεν θα τους πω τι να κάνουν. Αλλά βεβαίως γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία πρόθεση να φύγει από την Ευρωζώνη. Οι συνεχείς επαφές που έχουμε με τις ελληνικές αρχές, όχι μόνο με τις αρχές, με την αντιπολίτευση, ξέρουμε, οδηγούν στο να σας λέω ότι ξέρουμε πως δεν θέλουν να φύγουν από την Ευρωζώνη. Ίσως κάποιοι να θέλετε να φύγει η χώρα από την Ευρωζώνη ή να φύγει η δική σας χώρα από την Ευρωζώνη, αλλά δεν είναι η χώρα σας στην Ευρωζώνη, το σεβόμαστε. Η, η χώρα, η Ελλάδα, είναι αποφασιστικά μέσα στην Ευρωζώνη, έχει προβλήματα, αλλά δεν θέλει να φύγει. Η πραγματικότητα είναι, και το επαναλαμβάνω, ότι και χώρες εκτός Ευρωζώνης έχουν αντίστοιχα σχεδόν, τουλάχιστον αντίστοιχα προβλήματα. Η Ισλανδία δεν είναι στην Ευρωζώνη, αλλά πτώχευσε. Μία από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο πριν τη χρηματοοικονομική κρίση, κατά κεφαλήν. Στην Ένωση υπάρχουν χώρες που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα λόγω υψηλού επίπεδου δαπανών. Η πραγματικότητα είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι το ευρώ, αλλά το υψηλό επίπεδο χρέους ή ελλείμματος της οικονομίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που ήρθατε για μία ώρα ενώ μεταξύ μας απαντώντας σε πολύ δύσκολες μερικές φορές ερωτήσεις. Ευχαριστώ όλους σας. Ολοκληρώνεται η σχετική συζήτηση.